I'm honored to be... Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι στην Επιτροπή σα ω προτινόμενο επίτροπο για το φυλάκιο τη Διεθνού Συνεργασία και τη ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξωτερική δράση. Πρωταρχικό τη στόχο είναι να μειώσει και μακροπρόθεσμα να εξαλείψει την φτώχεια. Είναι μια πολιτική για τον κόσμο, για του πολίτε και ενισχύει την αλληλεγγύη, στηρίζεται σε αυτή γιατί είναι πυρήνας των ευρωπαϊκών αξιών αλληλεγγύη με του ανθρώπου που ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα και ρισκάρουν τη ζωή του για να φτάσουν σε ευρωπαϊκέ ακτέ με σχεδίε που και σαπιοκάραβα που συχνά γινόνται και τα θέρετρά του. Αλληλεγγύη προς τις γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλική βία ή ανθρώπου που διώκονται επειδή ανήκουν σε μειονότητε. Ε, αλληλεγγύη προς τα παιδιά στρατιώτες. Η αναπτυξιακή πολιτική αποσκοπεί στην εταιρική σχέση που στηρίζεται σε αμοιβέ συμφέροντα. Όταν ευάλωτα κράτη καταραίουν ή εξαπλώνεται η τρομοκρατία στην Αφρική, αυτό δημιουργεί άμεση απειλή για την Ευρώπη. Όταν αυξάνονται οι εμπορικέ ροέ και βελτιώνεται το κλίμα για τι επιχειρήσει, δημιουργούνται ευκαιρίες και για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταπληκτικέ επιδόσει στην αναπτυξιακή πολιτική. Μαζί με τα κράτη-μέλη αποτελεί το μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίω, προσφέροντας άνω του ίμιση του συνόλου της αναπτυξιακή βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρο των αναπτυσσομένων χωρών, καθώς και βασική πηγή τεχνολογίας, καινοτομία, επενδύσεων και επιχειρηματικότητα. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ε, ενίσχυσης και στην συνεκτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής αν, εγκριθώ, αν με εγκρίνετε ως Επίτροπο, δεσμεύομαι να αφιερώσω την εμπειρία μου και να, να προκειμένου να εξασφαλίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή, αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα έχει κέρια, ε, κέρια σημασία για το πρόγραμμα μετά το 2015 και τις διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο μετά τη διαδικασία Κοτονού και φυσικά για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής. Φτάνουμε στην πρώτη προτεραιότητα, ένα φιλόδοξο πλαίσιο μετά το 2015. Οι ισχύοντες αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας ε, απέφεραν ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενθαρρυντικά για τη μείωση τη ε, φτώχεια που έχει μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στο μισό. Σήμερα πολύ λιγότεροι άνθρωποι πηγαίνουν να κοιμηθούν νηστικοί, λιγότερα παιδιά πεθαίνουν από αρρώσει που μπορούμε να προλάβουμε και όλο και περισσότερα παιδιά, ιδιαίτερα κορίτσια, ε, παρακολουθούν ε, σπουδές. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα. Μία γυναίκα στην Αφρική έχει 29, 29 ε, περισσότερες 29 φορέ περισσότερες πιθανότητε να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Περίπου 750 εκατομμύρια στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλέ πόσιμο είδωρ. Και δυστυχώ ε, η φτώχεια είναι ακόμη μια συγκλονιστική πραγματικότητα. Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο πεθαίνουν από υποσυτισμό και λιμοκτονούν. Φυσικά υπάρχουν και αυξανόμενες ανισότητες και γεωγραφικά χάσματα. Και ενώ η Ασία και η Λατινική Αμερική βρίσκονται σε πιο καλό δρόμο, η υποσαχάριος Αφρική υστερεί. Πάνω από 120 εκατομμύρια διαβίουν σε απόλυτη φτώχεια, περισσότεροι από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Το πλαίσιο μετά το 2015 θα πρέπει να συμβάλλει στην εξάλληψη της φτώχειας και να συμβάλλει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να σταματούμε τη φτώχεια στη ρίζα της, το κακό στη ρίζα του. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση και να βρει την βέλτιστη ισορροπία μεταξύ τους. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου, καθώς και της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση να συνδυάσουμε όλες αυτές τις πτυχές και να τις εντάξουμε σε ένα ενιαίο οικουμενικό και περιεκτικό πλαίσιο που θα ισχύει για όλες τις χώρες τις πλούσιες και τις φτωχές. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ε, υλοποιήσουμε αυτή την πρόκληση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να διαμορφώσουν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και να αναλάβουν την ευθύνη το, της ανάπτυξής τους. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για κάποιον άλλον είναι όχι να μοιραστούμε τα πλούτη μας, αλλά να του δείξουμε ποιος είναι ο δικός του πλούτος. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας μετά το 2015 θα είναι η ανάπτυξη της χρηματοδότησης και κυρίως των μέσων εφαρμογής. Συμφωνώ πλήρως με τον, πρόεδρο, τον εκλεμμένο πρόεδρο Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στις, στους στόχους της χιλιετίας και να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να, να, να επενδύσουν τουλάχιστον 0,7% του ΑΕΠ τους στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το στόχο και να τον υλοποιήσουμε μέχρι το 2015, κάτι που προς το παρόν είναι ανέφικτο. Αναγνωρίζουμε βέβαια τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων χωρών της Ευρώπης, αλλά θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στα κρατη στο νέο πλαίσιο να τηρήσουν αυτή την υπόσχεση. Για να βελτιστοποιήσουμε την επίπτωση της ενίσχυσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο συντονισμό και στην ε, καλύτερο, καλύτερο συνδυασμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να αυξήσουν ε, τους εθνικούς τους πόρους ε, με χρηστή οικονομική διαχείριση, καλύτερη διακυβέρνηση, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και με αποτελεσματικά και δίκαια φορολογικά συστήματα. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάποια καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στην εξωπρεπή εργασία. Μόνο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, όπου όλοι οι συμβαλόμενοι θα παίζουν τον ρόλο τους, θα οδηγηθούμε στην επιτυχία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, προκειμένου να υιοθετήσει μια, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη συνολική ελληνική και την εξασφάλιση ενός αηφόρου μέλλοντος που δεν θα αποκλεί κανέναν. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να εγκαινιάσω και να διαπραγματευτώ ένα πλαίσιο για μετά τη Συμφωνία Κοτονού και μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική. Η υφιστάμενη Συμφωνία Κοτονού είναι η πιο περιεκτική συμφωνία βορρά-νότου στον κόσμο. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση. Βέβαια, οι χώρες ΑΚΕ είναι πολύ σημαντικές για μας περισσότερο από ποτέ θα έλεγα. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφώσουμε και θα σχεδιάσουμε καλύτερα τη συνεργασία μας στο μέλλον. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να αντικατοπτρίζει την έκβαση της διαδικασίας μετά το 2015. Δεν μπορεί να αποτελεί μια απλή συνέχιση του παρελθόντος. Η ομάδα των χωρών ΑΚΕ επίσης σκέφτεται την ε, συνέχεια της διαδικασίας και εμείς θα πρέπει το, να κάνουμε το ίδιο ενισχύοντας την εταιρική μας σχέση με τις χώρες ΑΚΕ φυσικά με βάση το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και λαμβάνοντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των χωρών και των περιφερειών. Θα πρέπει από κοινού να συζητήσουμε πώς θα προωθήσουμε την εταιρική μας σχέση. Ως πρώτο βήμα θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια ευρεία διαβούλευση και διάλογο τα επόμενα χρόνια. Η τρίτη μου προτεραιότητα είναι να συμβάλλω σε μια μεγαλύτερη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί ο κόσμος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ε, της ειρήνης, της ασφάλειας, της ενέργειας, των κλιματικών αλλαγών, της γεωργίας και του εμπορίου. Μεγαλύτερη συνοχή λοιπόν των εσωτερικών και εξωτερικών μας πολιτικών αποτελεί επιτακτική ανάγκη εκ των όνων προϋπόθεση και η συνεργασία που θα προσφέρουμε στους εταίρους μας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια αμυγή βοήθεια, αλλά να περιλαμβάνει θέματα όπως επιστήμη, υγεία, εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, νεολαία, εργασιακή κινητικότητα και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι θα πρέπει να περιλάβουμε νέα στοιχεία στο σχεδιασμό των πολιτικών μας. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ε, συνοχής των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η δομή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία στη, στην μεθοδολογία εργασίας με την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο, καθώς και τους υπόλοιπους επιτρόπους, θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας. Προσωπικά θα συμβάλλω στην υλοποίηση αυτών των προσπαθειών. Η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, την, πολιτική ανθρωπιστική βοήθειας, την εμπορική, την μεταναστευτική και άλλες πολιτικές. Αν εγκρίνεται ε, την... Αν με εγκρίνεται ως επίτροπο θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην συνοχή της ανάπτυξιακής πολιτικής και να έχω στενή συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Επίσης, θα παρακολουθώ την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών και θα έχουμε συνεργασία σε πρώιμο επίπεδο με τους υπόλοιπους επιτρόπους προκειμένου να προβούμε σε μία ενδελεχή ανάλυση των πρωτοβουλειών μας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμη ε, Ευρωβουλευτή κυρία Πρόεδρε, 83% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους, ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες. 61% των συμπολιτών μας πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια και 70% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η προσφορά ρογής σε αναπτυξόμενες χώρες έχει και για αυτούς θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής και να προβάλλουμε περισσότερο τα επιτεύγματά μας. Γι' αυτό και θα ήθελα μία πολιτική που να είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα και να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ. Το επόμενο έτος θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Θα είναι ιδανική ευκαιρία να έχουμε επαφή και διάλογο με τους πολίτες και να εξηγήσουμε πώς η αναπτυξιακή μας πολιτική είναι υποφελής για όλους μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, αν επιβεβαιώσετε την, το διορισμό μου, θα συνεχίσω να επιδιώκω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά θα τιμήσω τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο στρατηγικό και διορθωμένο διάλογο και θα επιδιώκω τακτικό και τακτικό άτυπο διάλογο μεταξύ μας. Τέτοιος διάλογος θα είναι πολύ σημαντικός ε, για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε ε, θετικά την διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού πλαισίου μετά το 2015 και να ε, αποφαινόμαστε με ενιαφωνή και να προασπίζουμε ένα ενιαίο όραμα. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτούς τους